Pan Przewodniczący! Good morning. Witam koleżanki, kolegów. Καλημέρα, καλώς ήρθατε όλοι. Συνεχίζεται η σύνοδός μας. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη η ε, έκθεση του κυρίου Βιταλκάδρας όσον αφορά τον ασφαλή αφοδιασμό με αέριο. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και πολλά χρόνια είδαμε σε πολλές περιπτώσεις την, το ευάλωτο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την παροχή ενέργειας και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της παροχής φυσικού αερίου το χειμώνα του 2005-2006 και 2008-2009 οι διακοπές εφοδιασμού στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν πραγματικά ένας εφιάλτης. Το γεγονό ότι ήταν σκληροί οι τελευταίοι χειμώνε στην Ευρώπη μα υποχρεώνει ακόμα περισσότερο να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να αποτρέψουμε παρόμοιε καταστάσει στο μέλλον η τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενέργεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από χώρε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά η διπλωματία μπορεί να επιτύχει πολλά σε αυτό το στρατηγικό τομέα. Έχουμε όλοι ε, ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό που ήταν αξιόλογες. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται να δημιουργήσουμε και μηχανισμούς οι οποίοι θα είναι πιο αποτελεσματικοί σε άμεσο επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι η κρίση εφοδιασμού με φυσικό αέριο, <clears throat> φυσικό αέριο που έχουμε αντιμετωπίσει οφείλονται στο ότι δεν υπήρξαν επαρκείς διασυνδέσεις και δεν υπήρξαν κατάλληλοι κανόνες αγοράς που να επιτρέψουν μια αλληλεγγύη αποτελεσματική μεταξύ των κρατών μελών. Ο κανονισμό τον οποίο θα ψηφίσουμε είναι ένα βήμα προς τα εμπρός για να επιληθούν τα προβλήματα αυτά. Είναι πολύ ο χρόνο που έχουμε δαπανίσει για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποια πρόοδο στον τομέα αυτό. Κατανοώ τι δυσκολίε οι οποίε προκύπτουν από τι διαφορετικέ εθνικέ ρυθμίσει και οι διαπραγματεύσει ήταν πολλέ φορέ εργώδει και δύσκολε. Αλλά η συμφωνία την οποία θα ψηφίσουμε τονίζει το ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να ξεπεράσουν τι ε, επιμέρου εθνικέ του θέσει για να καταλήξουν σε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στο σημαντικό αυτό πρόβλημα. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί αυτό ο κανονισμό. θα έχουμε στα χέρια μα ένα ισχυρό εργαλείο για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Ο κανονισμός αυτός ενεκρίθη στην Επιτροπή Βιομηχανίας Ενεργείας με ομοφωνία μετά από την ευτυχή κατάληξη των τριγωνικών διαλόγων με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω όλου του σκιώδες εισηγητέ για τη θαυμάσια εργασία και συνεργασία του μαζί μου, που τελικά αντανακλάται στο τελικό κείμενο, αλλά επίση και τα μέλη των εμπλεκομένων επιτροπών που γνωμοδότησαν προ την Επιτροπή Βιομηχανία και των οποίων τροπολογίε ενσωματώθηκαν στο κείμενο σε μεγάλο βαθμό. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την σημαντική της υποστήριξη προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και επίσης να αναγνωρίσω τη σημαντική συμβολή της Ισπανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο που μας κράτησε πάντα ενήμερο σε όλες τις χρονικές στιγμές για την κατάσταση των εργασιών του Συμβουλίου. Ο κανονισμός αυτός εξασφαλίζει την ασφάλεια όλων των πολιτών της Ευρώπης σε σχέση με τον εφοδιασμό σε ενέργεια. Από εδώ και πέρα θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και καλύτερα προστατευμένοι σε περίπτωση κρίσης. Και δίνει επίσης και κάποια ευελιξία στα κράτη-μέλη <clears throat> για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν πρόσθετους προστατευμένους πολίτες, ε, φορείς μάλλον, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες. Όταν ένα κράτος μέλος πρέπει να προστατεύσει την εθνική του αγορά και τους καταναλωτές, θα πρέπει να εξασφαλίσει μια ισορροπία σε ό,τι αφορά την παροχή ενέργειας βάσει της αρχής της αλληλεγγύης με τους πολίτες και των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός επιβάλλει την υποχρέωση στις επιχειρήσεις που παρέχουν φυσικό αέριο σε περίπτωση κρίσης να δώσουν κατά προτεραιότητα ε, φυσικό αέριο στους προστατευμένους πελάτες για ένα χρονικό διάστημα 30 ημερών χωρίς καμία διακοπή. Συγχρόνως όμως τα κρατημέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ή να ανανεώσουν τις δικές τους υποδομές ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ενσωμάτωση τη εσωτερική αγορά στην ενέργεια και να μην υπάρξουν <clears throat> νησίδες ενεργειακές μέσα σε εισαγωγικά. Ένας, μία από τις μεγάλες επιτεύξεις αυτού του κανονισμού είναι το ότι επιβλήθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη η δυνατότητα, η υποχρέωση μάλλον ανάδρομης ροής στις διασυνδέσεις φυσικού αερίου βασιζόμενη στις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται. Η ανάδρομη αυτή ροή θα επιτρέψει χάρη στις ε, επενδύσεις οι οποίες θα είναι περιορισμένες στον χρόνο και θα έχουν ε, κόστος το οποίο μπορεί να υπομειστεί κανείς μια σωστή κατανομή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Αυτό το βλέπουμε κυρίως και στον ε, ε, αγωγό που δίνει φυσικό αερίο στη Σλοβακία, Τσεχία και Πολωνία μέσω της Λευκορωσίας. Επίσης, η Κομισιόν αποκτά το δικαίωμα του ΒΕΤΟ σε σχέση με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία μπορεί να θεωρήσει ότι θέλουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε δύο λεπτά ακόμα στο τέλος της συζήτησης, λέει ο πρόεδρος, αν θέλετε. Σας ευχαριστώ. Και επίσης, η Κομισιόν θα ασκήσει με αποφασιστικό τρόπο τις εξουσίες της για το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών κατά τη διάρκεια κρίσεων μέσω της ομάδος συντονισμού για το φυσικό αέριο. Ο κανονισμός λοιπόν αυτός αποτελεί μια πραγματική λύση για ένα σημαντικό και απτό πρόβλημα, το πρόβλημα της ασφάλειας εφοδιασμού στην Ευρώπη και υποχρεώνει όλους τους φορείς της αγοράς να συνεργαστούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα προβλήματα τα οποία μπορούν να ανακύψουν σε σχέση με τον εφοδιασμό σε φυσική αέρια. Η σωστή και αποτελεσματική ε, παροχή αερίου στην αγορά. Η ενσωμάτωση καταναλωτών και παραγωγών και οι διασυνδέσει είναι η καλύτερη ασφάλεια έναντι των μελλοντικών κρίσεων. Κύριε Πρόεδρε, ο χαρισμό για την ασφάλεια σε εφοδιασμό φυσικού αερίου είναι ένα ποιοτικό άλμα, ένα σημαντικό ποιοτικό άλμα, βάσει του οποίου τα κράτη-μέλη εγκαταλείπουν τα καθαρά εθνικά συστήματά τους και μπαίνουν πλήρως σε ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχήμα. Είναι σίγουρο ότι ήταν απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις για να ε, κατανοήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και τα κράτη-μέλη ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των κρίσεων, αλλά σίγουρα διακόπτει, διακόπτει ο πρόεδρος. Κύριε Αντιπρόεδρε, είναι πολύ σημαντική. Κλείνω, κλείνω κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Βιδάλ Ο κανονισμός αυτός είναι ένα ιστορικό ορόσημο προς την ασφάλεια εφοδιασμού ευσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μία σημαντική απόδειξη της ε, πρόοδου που μπορεί να επιτευχθεί με το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή λοιπόν αυτού του κανονισμού θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους αυτούς οι οποίοι μας τροφοδοτούν με φυσικό αέριο που είναι πάντα σχεδόν φίλοι μα. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσουμε λέει ο πρόεδρος. Η Ευρώπη για όλους. Κύριε Αντιπρόεδρε, πάρα πολύ σημαντική η ομιλία, σημαντικότατη και η έκθεση. Ξέρω πόσο σημαντική είναι, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε σύμφωνα με τον κανονισμό. Χρησιμοποίησατε όλο τον χρόνο σας. Είχατε έξι λεπτά όλα μαζί, τώρα πήγατε στα 7 λεπτά. Στο τέλος δεν θα έχετε παρατηρήσεις κύριε Σιγητά και λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι. Εκ μέρους της ε, των, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γκίντερ Έτιγκερ. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βουλευτές, το φυσικό αέριο είναι ένα σημαντικός παράγον μέσα στην ενεργειακή μας πολιτική και ως εκ τούτου έχουμε καθήκον να εξασφαλίσουμε ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό χώρο σε ό,τι αφορά την παροχή φυσικού αερίου, να εξασφαλίσουμε επίση την ασφάλειά μα και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών από τι οποίε τροφοδοτούμεθα. Αυτό σημαίνει πρέπει να αναπτύξουμε την κατάλληλη υποδομή και συγχρόνω να ακολουθήσουμε μια κοινή γραμμή έναντι των εταίρων μα που παρέχουν ενέργεια και των χωρών διαμετακόμιση φυσικού αερίου. Έτσι λοιπόν θα μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά η αγορά φυσικού αερίου. Η κρίση του Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους, αλλά επίσης και η κρίση του Ιουνίου μεταξύ της ε, Ρωσίας και της Λευκορωσίας έδειξαν τη σημασία του φυσικού αερίου και της ασφάλειας ε, εφοδιασμού. Επί τη βάση της πρότασης της Κομισιόν λοιπόν έλαβαν χώρα οι διαπραγματεύσεις με, το κράτος μέλος, με τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο και μετά από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων κατέληξαν σε ένα επικοδομητικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα για την βιομηχανία και για τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδίω και προφανώς πάνω απ' όλα τον κύριο ε, Βιδάλ Κουάδρας για τον πολύ καλό τρόπο με τον οποίο μπόρεσε να διαιτητεύσει μεταξύ των διαφόρων απόψεων ώστε να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία θα ήταν αποδεκτή. Και επίση θέλω να ευχαριστήσω τα κράτη-μέλη που έδειξαν τη διαθεσιμότητα να εγκαταλείψουν εθνικέ αρμοδιότητε και να τι αφήσουν στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο αυτοκανονισμού είναι το πρώτο νομικό εργαλείο στα χέρια μα <clears throat> που μετά από τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας αντιμετωπίζει την ε, ε, εφαρμογή του άρθρου της συνήθειας Λισαβόνας για την ε, ενέργεια που δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέες ευρύτερες ε, αρμοδιότητες. Σε ό,τι αφορά τα θέματα λοιπόν ε, τροφοδοσίας με φυσικό αέριο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε αυτό το κοινό εργαλείο. Και πάλι πρέπει να τονίσω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του φυσικού αερίου ώστε <clears throat> να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια κοινή θέση στα θέματα της συμφωνίας της Πολωνίας με, την με τη Ρωσία που θα πρέπει να είναι σύμμορφη με τις με διατάξεις αυτού του κανονισμού. Θέλουμε επίσης να χαιρετήσουμε την αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κινηθούμε προς μια ευρωπαϊκή κοινή στάση στα θέματα αυτά βάσει των τεχνικών δυνατοτήτων όπως της ανάδρομης δρομής θα πρέπει να προχωρήσει η ανάπτυξη υποδομών ώστε να καταλήξουμε και σε μια κοινή πολιτική ενέργειας και επίσης και μια κοινή εξωτερική πολιτική ενέργειας. Είναι απαραίτητο επίσης να υπάρξει η εποπτεία της εσωτερικής αγοράς και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν ελάχιστες ελάχιστες προδιαγραφές. Αυτό είναι δείγμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και φροντίδας της Ευρώπης για τους πολίτες της. Επίσης όταν υπάρχουν ε, ακραίες συνθήκες θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να είναι απόλυτα δεσμευτικές σε στιγμές όπου είναι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή υπάρχουν εχμές ε, ζήτησης ενεργείας. Όλα αυτά δεν αποτελούν απλώς μαξιλαράκια, αλλά ε, διατάξεις οι οποίες θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την σωστή παροχή φυσικού αερίου, ιδίως στις δυσμενείς χειμερινές συνθήκες. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια ενιαία φωνή και προς τα μέσα και προς τα έξω και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την κοινή μας υποδομή στα θέματα αυτά. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει πολλά μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν για το θέμα των υποδομών. Η ανάδρομη ροή που αναφέρθηκε θα πρέπει να υποστηριχθεί με χρηματοδότηση και το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μιλών και εδώ αναφερόμαστε σε περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα πρέπει να δαπανηθούν ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτού του κανονισμού <clears throat> σε επίπεδο υποδομών. Παραμένουν πολλά τα οποία πρέπει να πράξουμε βέβαια και είμαι σίγουρος ότι αυτός ο κανονισμός δεν είναι η τελευταία λέξη στα θέματα της ενέργειας. Θα κάνουμε μια ενδιάμεση, μια ενδιάμεση αξιολόγηση στα μέσα του τρέχοντος έτους και στη συνέχεια θα δούμε σε, ποια, σε ποιους τομείς χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες. Ο στόχος μας είναι η ταχύτερη δυνατή εφαρμογή του κανονισμού από τη στιγμή που θα έχει εγκριθεί. Η Κομισιόν θέλει να είναι δραστήρια ιδιαίτερα για τα θέματα των εξωτερικών ενεργειακών σχέσεών μας επίσης. Έχουμε δημιουργήσει για το σκοπό αυτό μια ομάδα συντονισμού που βοηθάει την Κομισιόν η οποία θα βοηθήσει να δώσει στον κανονισμό αυτό ένα ενισχυμένο ρόλο. Χαιρετίζουμε το γεγονός αυτό ότι όχι μονάχα ε, στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες γύρω από την Ευρώπη θα μπορέσουν να εφαρμοστούν πιλωτικά προγράμματα του είδους αυτού. Δηλαδή ότι θα μπορέσουν να εξευρεθούν και περιφερειακές λύσεις μέσα στην σύνολη ευρωπαϊκή διάσταση και η Κομισιόν θέλει να υπάρξει μια ευρύτερη συζήτηση σε σχέση με το πακέτο υποδομών για τα θέματα ενέργειας, το οποίο θα παρουσιάσει τον Νοέμβριο και επίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά στην επόμενη περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο συνάδελφος Άρης Βόσκη δεν είναι παρόν. Εκ μέρους Επιτροπής Ένβη, Μπόγκουσλαβ Σόνικ. Έχετε το λόγο, συνάδελφε. Κύριο Σόνικ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για τους πολίτες, οι πολίτες Ευρώπης μάλλον περιμένουν σημαντικές αποφάσεις από την Ευρώπη. Θέλουν μια επίδειξη αλληλεγγύης. Θέλουν να μας βλέπουν να δρούμε σε διασυνοριακό επίπεδο. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτό που συζητούμε. Δηλαδή, δυνατότητα να υπάρχουν ε, μετακινήσεις διασυνοριακές για τους πολίτες Ευρώπης. Είναι και θέμα ασφαλούς εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Επί έτη κάναμε εκστρατεία για, για τον ασφαλή εφοδιασμό σε φυσικό αέριο και να θεωρηθεί προτεραιότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να εξαρτώμεθα μόνο από έναν προμηθευτή φυσικού αερίου, δηλαδή από τη Ρωσία. Η Ρωσία χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο σαν ένα μοχλό ασκήσεως πιέσεως επάνω μας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε όλους ιδιαίτερο το θέμα. Εμείς ως Πολωνοί αναφερόμαστε στο πρόγραμμα North Stream το οποίο ήταν ένα έργο που αποφασίστηκε χωρίς σωστή διαβούλευση με τις χώρες ε, που ενδιαφέρει άμεσα το θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, το οποίο σύστημα θα εγγυάται τον ασφαλή εφοδιασμό σε φυσικό αέριο για κάθε κράτο μέσω Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρο. Η κυρία Σάντρα Καλνιέτε έχει το λόγο. Επιτροπή ΙΜΚΟ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ σημαντική είναι αυτή η έκθεση. Και χαίρομαι που το ψήφισμα του Κοινοβουλίου αντικατοπτρίζει τον φόβο των χωρών μελών εκείνων που είναι απομονωμένε όσον αφορά την ενέργεια, διότι εξαρτώνται κυρίως από εφοδιασμό από τρίτε χώρες και δεν έχουν αρκετές διασυνδέσει με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, ελπίζω ότι αυτός ο κανονισμός θα μας βοηθήσει, θα βοηθήσει να αναπτύξουμε έναν χώρο, έναν τομέα ε, ενεργειακού εφοδιασμού κοινό, σαν μέλος Επιτροπής ΣΥΜΚΟ, Εκτιμώ διάφορε βελτιώσει που επέφερε το Κοινοβούλιο στην πρόταση. Πρώτα απ' όλα, είναι πιο ακριβή ο ορισμός των προστατευμένων πελατών που σε δύσκολε περιστάσει εφοδιάζονται σε φυσικό αέριο. Δεύτερον, έχουμε ενισχύσει και την αρχή τη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκή Ενώσεω, υπογραμμίζοντας την συνεργασία μεταξύ περιφερειών και αυξάνοντας τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τέλος, αναφερόμενοι στι διακοπές εφοδιασμού, η προτεραιότητα δίδεται στα μέσα τη αγορά και όχι στα εξωτερικά μέτρα εκτός αγοράς που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις εκείνες κατά τι οποίε η αγορά δεν μπορεί να εξασφαλίζει τον ασφαλή εφοδιασμό των προστατευμένων πελατών. Και τέλο, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βιλακουάδρα για την έξοχη συνεργασία μα. Η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική, λέει ο Πρόεδρο, αλλά παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σα. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Ο συνάδελφο Αρεσβόλσκι ε, από την Επιτροπή ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο ασφαλή εφοδιασμό ενέργεια είναι βασικό στοιχείο για τη διαφύλαξη του μέλλοντος και είναι καλό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να παρέχει αυτό το αγαθό μάλλον στους πολίτες της. Το θέμα δεν είναι εάν, αλλά πώς θα πρέπει να δράει η κοινότητα, τόσο ότι τα κράτη-μέλη να είναι ασφαλή όσον αφορά τον εφοδιασμό σε ενέργεια. Γι' αυτό χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υπάρχει το σωστό νομοθετικό μέσο και δεύτερον χρειάζεται ένα πολιτικό όραμα και η προθυμία να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Τόσο αφορά το νομοθετικό πακέτο το οποίο διαπραγματευθήκαμε με αποτελεσματικό τρόπο και διαπραγματεύτηκε πολύ αποτελεσματικά και ο ο στόχο είναι ασφαλή εφοδιασμό ενέργεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι κατά δύο τρίτα έχει επιτευχθεί ο στόχο εν συγκρίση με τι αρχικέ φιλοδοξίε που είχαμε θέσει. Μα παρέχει φιλόδοξου κανόνε όσον αφορά τι υποδομέ, εισάγει ένα σύστημα κοινωνική αντίδραση σε κατεπίγουσε περιπτώσει, συμπεριλαμβάνει στο άρθρο 104 την αρχή τη αλληλεγγύη τη συνθήκη, που είναι στο άρθρο 104 τη συνθήκη. Υπάρχουν όμω και παραλήψει σημαντικέ, κυρίω όσον αφορά την εξωτερική διάσταση τη ενεργειακή πολιτική Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ο κανονισμό δεν αναφέρεται στον ρόλο τη ΥΠΑ τη και μόνο όριστα αναφέρεται στο νότιο διάδρομο ή Ναμπούκο και τη συνεργασία με άλλου μα εταίρου. Το κείμενο εν γέννη είναι τεράστια πρόοδο. Εάν εφαρμοστεί σωστά θα είναι μεγάλη πρόοδο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Ευχαριστώ διακόπτη ο Πρόεδρο. Χρειάζεται αλληλεγγύη τα κάτι μελη να μπορούν να αποφασίσουν ποια θα είναι η δομή του εφοδιασμού του φυσικού αέριο. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω συμπερίληψη. Λυπάμαι, διακόπτη ο Πρόεδρο. Τέλο του χρόνου σα. Τέλο χρόνου. Ένα λεπτό είχατε. Συνεχίζει ο κ. Σαριουσβόλσκι και διακόπτει και το μικροφόνο του. Λοιπόν, συνάδελφοι, ο Πρόεδρο, παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σα, διότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε κανονικά στι εργασίε μα. Για όλους ισχύει το ίδιο. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν. Εκ μέρους του ΕΛΚ. Herbal Royal. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω ε, εν θέρμος όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν εργαστεί στα πλαίσια αυτού του εγχειρήματο, ιδίως τον κύριο Βιδάλ Κουάδρας. Αυτό απέδειξε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική είναι σε θέση να αντιμετωπίζει κρίσεις και να παρέχει λύσεις που θα εμποδίσουν την επανεμφάνιση αυτών των κρίσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ε, ασφάλειας ευωδιασμού. Υποχρεωθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και το έχουμε αντιμετωπίσει. Βρήκαμε λύσεις οι οποίες δεν ήταν εύκολες, δεν ήταν απλές, οι οποίες απίτησαν και τη δημιουργία νέων εργαλείων και αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί δεν σημαίνει μονάχα νέα πρότυπα για τις υποδομές, αλλά και κοινού κανόνε για την πρόληψη κρίσεων στο μέλλον. Και όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Επίτροπος, αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα εξασφαλίσουμε 30 μέρες ασφάλειας εφοδιασμού για τους προστατευμένους ε, πολίτες. Αλλά και φορείς. Αυτό όμως κατέδειξε επίσης ότι είμαστε σε θέση να προβούμε σε συμβαστικές λύσεις, οι οποίες οδηγούν σε ληστελείς αποφάσεις σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων. Με τον τρόπο αυτό φυσικά παίζει κάποιο ε, τονίζεται και η ευθύνη των επιχειρήσεων που είναι υποχρεωμένες να εξασφαλίζουν τη διασύνδεση των υποδομών αλλά επίσης είναι σωστό να τονίσουμε ότι με τον τρόπο αυτό δεν πρέπει να υποχρεώσουμε κανένα σε ένα στενό κορσέ που δεν ξέρουμε πού θα μα οδηγήσει. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία, πρέπει να υπάρχει ανάδρομη δρομή, αλλά αυτό εξαρτάται πάντα από τι καταστάσει αγορά και τι τιμέ. Επομένω, αυτό μα δίνει μια μεγαλύτερη ευελιξία και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο και αυτό καταδεικνύει ότι και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν το δικό του μερίδιο ευθύνη. Όταν όμω δεν μπορεί να υπάρξει λύση από τα κράτη-μέλη, θα πρέπει τελικά η Κομισιόν να αποφασίσει σε τελική ανάλυση, μια κομισιόν η οποία είναι πολύ πιο ενισχυμένη για τα θέματα αυτά, η οποία θα πρέπει να έχει το τελικό λόγο αν δεν μπορούν να επικρατήσουν άλλες λύσεις. Λοιπόν, μιλάμε για μεγαλύτερη ευελιξία σε κατανομή βαρών στις περιπτώσεις κρίσεων. Υπάρχει λοιπόν ένα σύνολο λύσεων που έρχονται από τις Βρυξέλλες και για μια φορά είναι πολύ θετικές για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ήταν η πρώτη ομιλία που δεν ξεπέρασε το χρόνο της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Χέρπερτ. Ο συνάδελφος Χάν Σφόμποντα, αντιπρόεδρος, Σοσιαλιστικής και δημοκράτες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ φυσικά θα πρέπει να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Βιδάλ Κουάδρας για την πολύ καλή εργασία του, την έκθεσή του και φυσικά και με την, για την αγαστή του συνεργασία με όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Και όπως ανέφερε ήταν σημαντικός και ο ρόλος της Ισπανικής Προεδρίας. Ο κανονισμός αυτός αφορά την αλληλεγγύη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το κέντρο, το οδηγό νήμα της έκθεσης αυτής για το φυσικό αέριο, αλλά επίσης και η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Ορισμένοι θεώρησαν ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο είναι ε, αξίζει επικρίσεις, εμείς θεωρήσαμε ότι πρέπει να δώσουμε αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα προς τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους υποστηρίξουμε. Πρόσφατα εξεδόθη η έκθεση από την ομάδα του Jacques Delors για τη δυνατότητα να έχουμε μια ευρωπαϊκή διάσταση στα θέματα ενέργειας και ξέρω ότι και ο πρόεδρο μα έχει υποστηρίξει ιδιαίτερα αυτό το σημείο γιατί για μένα νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της πρόοδου της διαδικασίας ολοκλήρωσης Ευρωπαϊκό Ένωση. Τώρα μπορούμε να έχουμε μια κοινή πολιτική ενέργεια στα πολιτική συγγνώμη, Ευρωπαϊκή πολιτική στα ενεργειακά θέματα, χωρί να υπάρξει και τροποποίηση των συνδικών. Δεν πρέπει να εμπλακούμε σε μια συζήτηση για τροποποίηση των συνδικών. Είναι απαραίτητο όμω η αλληλεγγύη να τεθεί στο προσκήνιο να υπάρξει μια κοινή δράση και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το εσωτερικό είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε πολύ περισσότερες υποδομές, όπως τόνισε ο κύριος Επίτροπος, και πρέπει επίσης να δώσουμε και μεγαλύτερη έμφαση στις ανανεώσιμες ενέργειες, στην ηλιακή και την αιωλική ενέργεια. Αν μπορέσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη ικανότητα <clears throat> αποθήκευσης ενέργειας, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις κρίσεις γιατί θα μπορούμε να αντικαταστήσουμε την έλλειψη ενέργειας από φυσικό αέριο με άλλες ε, ενέργειες, με μορφές ενέργειας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αναπτύξουμε αυτές τις υποδομές. Έχουμε μια αγορά που είναι όλο και πιο κοινή. Άλλες χώρες όπως η Ρωσία δεν έχουν όμως ε, ε, ανοιχτή και ενιαία αγορά, έχουν μονοπωλιακές δομές και πρέπει να έχουμε ένα κοινό τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τις χώρες αυτές που είναι προμηθεύτριες μας. Πρέπει λοιπόν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αερίου στο μέλλον και αυτές να εξασφαλίσουν μια κοινή δράση που θα οδηγήσει σε καλύτερα τιμολόγια για τους ε, καταναλωτές και τους πολίτες. Λοιπόν, αυτό είναι μια πρόοδος η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε καλύτερα με το χρόνο τώρα. Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας. Η κυρία Μπαλεάννα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βιντάλ Κουάντρας για τη θαυμάσια δουλειά που έκανε για αυτή τη σημαντική έκθεση. Ο βαρύς χειμώνας μας θυμίζει πόσο εξαρτώμεθα από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Η ασφάλεια της παροχής ενέργειας είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι καλό πράγμα αυτό. Θέλουμε να μειώσουμε το ευάλωτο της Ευρώπης ώστε οι πολίτες να ξέρουν ότι παρά τη διαταραχή που ενδεχομένω θα υπάρξει θα έχουν παροχή αερίου. Αλλά χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές εφοδιασμού. Η ασφάλεια του εφοδιασμού είναι διαφορετική, έχει διαφορετικό νόημα ανάλογα με το πολίτης ποιας χώρας είστε. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή προσέγγιση όμως και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμπληρώσουμε σωστά την ενεργειακή αγορά. Έχουμε πολλά προστατευτικά εμπόδια παρόλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εξακολουθούν οι τιμές να είναι υψηλέ και υπονομεύεται η ο εφοδιασμός. Η πολιτική ε, ε, πολλοί λένε ότι οι πολιτικοί δεν πρέπει να ασχολούνται με την ενέργεια αλλά κάθε μέρα ακούμε για κλειστές πόρτες και συμβόλαια από τα οποία υπογράφονται στη Ρουμανία η στρατηγική μας η ενεργειακή είναι στα χέρια ολίγων και στα χέρια του Συμβουλίου Ασφαλείας που ε, προεδρεύει ο πρόεδρος οι συνέπειες αυτές της πολιτικής όμως ε, είναι στα χέρια των πολιτών όταν παίρνουν το λογαριασμό στο τέλος του έτους. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια, δημοκρατία και υπευθυνότητα από όλου αυτού που ασχολούνται με την ενεργειακή πολιτική. Αλλιώ δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση των καταναλωτών. Η ελεύθερη αγορά σίγουρα θα ρυθμίσει καλύτερα τα πράγματα από του πολιτικού. Θέλουμε λοιπόν η Κομισιό να καταργήσει τα εμπόδια, τα προστατευτικά. Ευχαριστώ κυρία μου. Εκ μέρους των Πρασίνων, ο Κλωτ Τούρνες, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ όλους αυτούς από εμά οι οποίοι έλαβαν μέρος στην επεξεργασία και τη διαπραγμάτευση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ και την Ισπανική Προεδρία η οποία προώθησε αυτό το θέμα μέσα σε στενά χρονικά θέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το θέμα για την καλύτερη σχεδίαση της ενεργειακής τροφοδοσίας μέσα στην Ευρώπη και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και χαίρομαι πολύ που έχει περάσει και η, η, έννοια της ανάδρομης ροής η οποία επιτρέπει μια μεγαλύτερη ευελιξία. Θέλω απλώ να αναφερθώ ότι στο γεγονός ότι στα θέματα των υποδομών είναι απαραίτητο να υπάρξουν και εγκάρσιες διασυνδέσεις, δηλαδή προς τα νότια και βόρεια, από την Πολωνία προς Σλοβακία και Ρουμανία. Και επίσης το θέμα που ανέφερε ο κύριος ε, ε, Σβόμποντα. Το θέμα της αποθήκευσης. Όταν υπάρχει περισσότερο φυσικό αέριο από ό,τι χρειάζομαι, από ό,τι χρειαζόμαστε στους αγωγούς, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης. Να υπάρχει λοιπόν αποθήκευση η οποία μπορεί να είναι μακροχρόνια μεν, αλλά να αποδίδει φυσικό αέριο στην κατανάλωση ταχαίως όταν αυτό είναι απαραίτητο. Δεύτερον, κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο ελείπει από τον τωρινό κανονισμό είναι η ικανότητα να έχουμε τα δεδομένα τα οποία θα μας επιτρέψουν να προβλέψουν τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> Ποιες θα είναι οι ανάγκες της αγωγής φυσικού αερίου στην ε, Γερμανία παραγωγικά το 2015 όλα τα, όταν όλα τα κτίρια μας θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια καλύτερη σχεδίαση στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν τα δεδομένα τα οποία θα μα επιτρέψουν να κατευθύνουμε καλύτερα και τι επενδύσει στον ενεργειακό τομέα. Τρίτον, στις 4 Φεβρουαρίου θα γίνει κάποια συνάντηση των αρχηγών κρατών για τα θέματα ενέργειας. Αλλά η Κομισιόν θα πρέπει προηγουμένως να έχει μια καλύτερη ε, ακτίμηση <clears throat> ε, της παγκόσμιας αγοράς ε, στον κόσμο. Οι ασβεστολιθικοί σχιστόλιθοι στι ΗΠΑ και στον Καναδά έχουν απελευθερώσει περισσότερη δυνατότητα φυσικού αερίου. Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη, τι κάνουμε στην Ευρώπη με αντίστοιχα πετρώματα, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε εμεί να έχουμε μια καλύτερη αξιολόγηση τη ενεργειακή πραγματικότητα από ό,τι πριν από τρία-τέσσερα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, ο συνάδελφο Σιμάνσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά. Πρέπει να σας συγχαρώ, κύριε Βιντάλ Κουάντρας. Πραγματικά καταφέρατε να βρείτε ένα συμβιβασμό. Αλλά ταυτόχρονα πετύχατε και σπάνια συνένεση μέσα στο πλαίσιο του Ευρωκοινοβουλίου. Η ομάδα των μεταρρυθμιστών είναι υπέρ αυτού του κειμένου. Έστω και αν στην αρχή ξεκινήσαμε να υποστηρίζουμε ένα πιο φιλόδοξο κείμενο όσον αφορά τις υποδομές και τις δεσμεύσεις σε περίπτωση κρίσης και σχετικά βέβαια και με τη διεθνή πτυχή της υπόθεσης. Πρέπει να σας πω ότι η πρώτη έκδοση του κειμένου ήταν πιο δεσμευτική και για τις επιχειρήσεις και για τα κράτη. Σήμερα ε, το κείμενο εμπεριέχει ακόμη ορισμένες δυνατότητες, αλλά ελπίζω ότι αυτό δεν θα αποτελέσει πρόσχημα για να συνεχίσουμε τη σημερινή μας πολιτική η οποία βασικά είναι μια πολιτική αδιαφορίας προς τη Ρωσία που χρησιμοποιεί το αέριο σαν πολιτικό μέσο στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης. Ελπίζω ότι θα καταπολεμήσουμε το μονοπόλιο της Gazprom. Για πολιτικούς λόγους θέλουν να διατηρήσουν τον πλήρη έλεγχο ε, στους αγωγούς αερίου στην Ευρώπη και ακόμη θέλουν και τον έλεγχο των πρώτων υλών δηλαδή μετά την πώληση του αερίου. Αυτό ε, απομειώνει τα δικαιώματα των πολιτών και υπονομεύει τις νέες τεχνολογίες στον χώρο του αερίου. Η έκθεση αυτή μας δίνει μια ευκαιρία και μια εγγύηση για μια ενιαία πολιτική εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσάκη Έναν. εκ μέρους της Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια ε, του εφοδιασμού, ναι, και την ανεξαρτησία, ναι, αλλά για να τα πετύχουμε αυτά πρέπει να αφαιρέσουμε το αέριο και τις άλλες ενεργειακές πηγές από την κερδοσκοπία. Πρέπει να έχουμε δασμολογικές συμφωνίες με τις χώρες παραγωγούς, παραγωγής, εξασφαλίζοντας τον πολίτη της Ευρώπης θα μπορούσε να είναι η αποστολή ενός Ευρωπαϊκού Φορέα Ενέργειας κάτω από τον ελεγχό μας. Δεν πρέπει να είμαστε στα χέρια των πολιεθνικών, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφές που αντιμετωπίσαμε στις, έξω από τις ακτές της Φλόριδας. Όλα αυτά εξυπηρετούν μόνο τους μετόχους των πολυεθνικών ενώ δεν δίνουν τη δυνατότητα στις χώρες παραγωγής να διαθέτουν ελεύθερα ε, το προϊόν τους. Ακόμη πιστεύω ότι η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού. Πρέπει να κρατικοποιηθεί κρατικοποιήσουμε στην Ευρώπη όλες αυτές τις επιχειρήσεις και να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό όμιλο κάτω από δημόσιο έλεγχο. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Η κυρία Νίκη Τζαβέλα. Κύριε Κουάδρας, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική αναφορά η οποία βάζει σε σειρά, σε μια τάξη, την εσωτερική μας αγορά θα ήθελα όμως να ξεκαθαρίσω το εξής κυρίες και κύριοι ότι σε καμία περίπτωση η ευρώπη δεν έχει διασφαλίσει δεν έχει λύσει το μεγάλο της πρόβλημα που είναι οι εναλλακτικοί προμηθευτές αερίου. αντιθέτως κύριε επίτροπε θα έλεγα ότι αν παρακολουθήσει κανείς ποιοι είναι οι προμηθευτές για την βιωσιμότητα των αγωγών αερίου που έχουμε σχεδιάσει ως ευρώπη θα δείτε ότι παραμένει ο ένας και μόνος προμηθευτής. η ρωσία έχει διασφαλίσει συμφωνίες προμήθειας αερίου με κάθε δυνατό προμηθευτή της ευρώπης ακόμα και με το ιράν για να φανταστείτε πόσο κυκλικά και ωραία μας έχει περικυκλώσει. δεν έχω αντίρρηση. σε αυτή την περίπτωση κύριε επίτροπε θα έπρεπε να δείτε με τον κύριο ταγιάννη να βρούμε μια αμοιβαία πρόταση εμπορικών δεσμεύσεων της ρωσίας προς αυτή την κατεύθυνση για να μπορούμε και εμείς να δεσμεύσουμε οικονομικά τη ρωσία. και σας ερωτώ ένα θέμα έχετε σκεφτεί δεν βλέπω να επιταχύνεται το action plan για το lng προμηθευτές από βόρειο αφρική και από τον κόλπο υπάρχουν προτίθεστε να αυξήσετε τα lng terminal στη μεσόγειο; εναλλακτικοί προμηθευτέ υπάρχουν κύριε επίτροπε και σας παρακαλώ να το προσέξετε. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία μου για τα σχόλιά σας. Ο συνάδελφος Μπέλα Κόβατς. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μιλάμε για μια σφαιρική αγορά αερίου. Το γεγονός ότι έχουμε εθνικοποιήσει ορισμένα στοιχεία. Αυτό μας οδήγησε σε συγκρούσεις με επιπτώσεις άμεσες ή έμεσες στην αγορά. Διαταράσει δυστυχώς τον εφοδιασμό οποιοδήποτε σχήμα για την παροχή αερίου μόνο μεσοπρόθεσμα μπορεί να αντιμετωπίσει τις τεχνολογικές ανανεώσεις και τον εφοδιασμό. Δεν μπορεί να προχωρήσει σε ευρύτερη διάσταση και δεν μπορεί πραγματικά να λάβει υπόψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Πρέπει να έχουμε ασφάλεια της προμήθειας, πρέπει να είναι εγγυημένη. Ο εφοδιασμός πρέπει να είναι σταθερός για τους καταναλωτές ε, σε τιμή λογική. Η ασφάλεια λοιπόν του εφοδιασμού και είναι σημαντική και η πολιτική αυτή είναι σημαντική για όλους μας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζουμε τα σωστά μέτρα για να προμηθεύουμε σωστά τα νοικοκυριά. Δεν μπορούν να αγωνιστούν τα νοικοκυριά για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Σήμερα έχουμε ελεύθερη αγορά αερίου. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος και οι άλλες αρχές πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα. Σας ευχαριστώ για την ομιλία σας. Ήταν συντομότερη από τον διαθέσιμο χρόνο μάλιστα. Για επόμενοι ομιλητές. Ο κύριος Κάριντς, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όλοι εξαρτώμεθα, όλοι εξαρτώμεθα στην Ευρώπη από τον εφοδιασμό από τρίτες χώρες ως προς την ενέργεια. Και είμαστε ιδιαίτερα εξερθυμένοι όσον αφορά το αέριο. Και η έντονη εξάρτησή μας ε, προκύπτει από τη Ρωσία. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, η Ρωσία σαν προμηθευτής μπορεί να είναι προβληματική χώρα. Το 2009 ο καυγάς μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας δημιούργησε μια κατάσταση που σήμαινε ότι πολλά κρατημέλη μείνανε από αέριο. Τώρα μπορεί να υπάρξουν δύο λύσεις. Η πρώτη είναι η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού. Η άλλη είναι η διασύνδεση της εσωτερικής αγοράς. Αυτά είναι λοιπόν που συζητάμε τώρα. Την κοινή ενεργειακή μας πολιτική. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια λειτουργική κοινή αγορά. Πού προκύπτει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλές χώρες και πολλές περιφέρειες στην Ευρώπη που είναι τελείως απομονωμένες από τις υπόλοιπες. Οι βαλτικές χώρες 100% απομονωμένες, 100% εξαρτημένες από τον εφοδιασμό από τη Ρωσία. Και το αποτέλεσμα είναι ότι στις βαλτικές χώρες σήμερα οι καταναλωτές πληρώνουν 30% περισσότερο για το φυσικό αέριο από ό,τι στη Γερμανία. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτός ο κανονισμός ακολουθεί την σωστή κατεύθυνση αυτά τα οποία έπραξαν η Κομισιόν και ο κύριος Κουάντρας μας οδηγούν στη σωστή τροχιά. Αλλά πρέπει να φτάσουμε και στο τέλος, στο στόχο. Δηλαδή χρειαζόμαστε επενδύσεις για υποδομές ώστε να έχουμε μια κοινή αγορά στον ενεργειακό τομέα για να μπορέσουμε να έχουμε πολλές πηγές προμήθειας και ασφάλεια. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, η κυρία Τερέζα Ριέρα Μαντουρέλ. Ένα λεπτό μόνο έχετε κυρία μου, λυπάμαι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αναφέρθηκε ήδη σήμερα η σημασία της κρίσης του 2009, η οποία έκανε ανάγλυφο, κάτι το οποίο δεν είχαμε συνειδητοποιήσει απόλυτα μέχρι τότε, ήταν η ενεργειακή μας εξάρτηση. Καταλάβουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος ήταν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ισπανία, παραδείγματος χάρη, δεν μπόρεσε να βοηθήσει τα εννέα κατημέλη τα οποία α, ε, επλήγησαν, διότι δεν είχε τους απαραίτητους πόρους για κάτι τέτοιο. Παρά το γεγονός ότι φαίνεται προφανές, η εσωτερική αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί τη δυνατότητα ταχεία μετακίνηση φυσικού αερίου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί συμβατικά ή τεχνικά ε, εμπόδια μέσω διαμεθοριακών διασυνδέσεων που σήμερα πόρο απέχουν από το να υπάρχουν σε επαρκέ επίπεδο. Εξού και η σημασία αυτού του κανονισμού που με τρόπο σαφή συνδέει την δημιουργία διασυνδέσεων στην, με την ασφάλεια εφοδιασμού και βασίζεται επομένω στην ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη διαφοροποίηση των ενεργειακών μα πηγών και να μπορέσουμε να καταργήσουμε, να ε, ξεπεράσουμε τις ενεργειακές νησίδες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και την Κομισιόν και τον κύριο Βιδαλκουάδα ως εισηγητή, αλλά και την Ισπανική Προεδρία που έχουν σε χρόνο ρεκόρ συμβάλει στο να μπορέσει να υλοποιηθεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και στον τομέα της ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία μου για την ομιλία σας. Διακόπτει ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριο Χατζημαρκάκη τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Έτιγκερ, τον Επίτροπο και τον κύριο Βιδάλ Καουάντρα για την έκθεσή του, ο οποίο επίση και με την, είχε την αρρωγή τη Ισπανική Προεδρία. ήταν μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Το φυσικό αέριο είναι σημαντικό, το τόνισε και ο κλάουτ Τόρμε. Θα γίνει πιο σημαντικό στο μέλλον. Θα πρέπει να αλλάξουμε την εξάρτηση αυτή η οποία φτάνει το 40% από την Ρωσία σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν σωστό και σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε τα απαραίτητα σχέδια πρόληψη για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες κρίσεις σε τρία επίπεδα πρόληψης για να αποφύγουμε την κρίση του 2001 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος μας είναι να έχουμε ευρωπαϊκές χώρες εταίρους, αλλά όχι εταίρους που μας αφήνουν στα κρύα του λουτρού ή στα κρύα του χειμώνα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε μια υπευθυνότητα όχι μόνο για τα κράτη-μέλη μα, αλλά και για χώρε οι οποίε είναι όμορε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλή η νόμη, κυρίε και κύριοι, χρειαζόμαστε και άλλου τρόπου να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Γι' αυτό χαιρετίζω την πρόταση του κυρίου Ρέτεγκερ να δώσουμε μία έμφαση σε περαιτέρω Μορφέ υποδομών όπω είναι το South Stream και το Ναμπούκο ώστε να μην εξαρτώμαστε από μία μονάχα πηγή τροφοδοσία σε φυσικό αέριο και επίση χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη ικανότητα αποθήκευση. Στην Γερμανία έχουμε μονάχα 70 ε, ημέρε αποθήκευση φυσικού αερίου δεν είναι απαρκέ. Θα πρέπει να έχουμε αρκετή αποθήκευση ενέργεια για να καλύψουμε την ανάγκη και των γειτονικών χωρών και αυτό πρέπει να εξασφαλίσει διαφοροποίηση και των πηγών τροφοδοσία σε φυσικό αερίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Τσοκανόφσκι, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρώπη είχε ένα πρόβλημα με τη διαταραχή του εφοδιασμού από τη Ρωσία. Την αποκαλέσαμε κρίση του αερίου τον Ιανουάριο του 2009. Να είμαστε προσεκτικοί όμως, διότι αυτό δεν επηρέασε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανάλυση κατέδειξε ότι επρόκειτο για διαρθρωτικό πρόβλημα αντί για κάτι άλλο. Λοιπόν, γι' αυτό χρειαζόμαστε να είμαστε περισσότερο ευαίσθητοι εδώ, να μην αναζητούμε περισσότερες ρυθμιστικές διατάξεις από όσες απαιτούνται, γιατί η υπερρύθμιση του εφοδιασμού μπορεί να αυξήσει τις τιμές του αερίου και να οδηγήσει σε περίπλοκες καταστάσεις για τους καταναλωτές και να καταργήσει και την, τον ανταγωνισμό. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η έκθεση κατάφερε να πετύχει μια σωστή υπηρεσία, μια λογική λύση. Και συμφωνώ με τον Επίτροπο ότι χρειάζεται μια αναθεώρηση αργότερα για να δούμε τα αποτελέσματα των μέτρων. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Ράντσορφ δεν είναι μαζί μας. Ο κύριος Φιωρέλο Προβέρα. Ένα λεπτό έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή παραγωγή φυσικού αερίου συνεχώς ε, μειούται και η ζήτηση ενεργειακή θα αυξηθεί κυρίως ε, στο εγγύς μέλλον ανάλογα με την οικονομική ανάπτυξη που όλοι περιμένουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν εφαρμόσουμε πολιτικές εφοδιασμού και σίγουρου και αυθόνου κυρίως σε περιπτώσεις κρίσεων όταν ο εφοδιασμός φυσικού αερίου εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες γεωπολιτικού. Αυτός ο κανονισμός βελτιώνει κατά πολύ τον συντονισμό μεταξύ των φορέων του τομέα του φυσικού αερίου και θα εμποδίσει να επαναληφθούν καταστάσεις όπως αυτή της κρίσης μεταξύ Ρωσία και Ουκρανίας χωρίς όμως να αμφισβητούνται τα προνόμια κάθε κράτου μέλους στο ενεργειακό πεδίο. Συγχαίρω τον εισηγητή, τον κύριο Βιδάλ Κουάδρας και τον ευχαριστώ που έλαβε υπόψη του κάποιες από τις τροπολογίες μας που είναι πολύ σημαντικές για μας. Ε, με χαρά άκουσα και αυτά που είπε ο Επίτροπος που θέλει να έχουμε καλύτερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά τον τομέα αυτό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκ Γκρίφιθ, Γκρίφιν, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρο, οι νομικοί κυνηγάνε τα νοσοκομιακά όπου υπάρχει ατύχημα, υπάρχει ένα παράσιτο που τρέχει για να βγάλει κέρδη από το ατύχημα κάποιου αλουνού που είναι υπέρ τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθούν κατεξοχήν τα νοσοκομιακά από τους σεισμούς, ε, πυρκαγιέ σε δάση, αύξηση θερμοκρασία. Κάθε κρίση γίνεται δικαιολογία για να αρπάξουν περισσότερες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση Ρωσία και Ουκρανίας ήταν τεχνητό πρόβλημα που δημιουργήθηκε από κάποιες παρεμβάσει οικονομικέ στην Ανατολική Ευρώπη. Η απάντηση είναι να σταματήσουμε αυτά και τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνουν ελεύθερα και να αγοράσουν το αέριο που θέλει να πουλήσει η Ρωσία. Αντί αυτού, η κρίση χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αρπάξει τον έλεγχο του εφοδιασμού φυσικού αερίου και να παγιδευτούμε όλοι σε μια αλληλεξάρτηση που θα υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάτι που ποτέ δεν θα ανέκριναν οι ψηφοφόροι. Δεν είναι θέμα εφοδιασμού σε ψηφικό αέριο, είναι η τυραννία ενό ε, σοσιαλιστικού υπερκράτου που προσπαθεί να αρπάξει με κόλπα αυτά που δεν παραπάξει δημοκρατικά. Όταν λοιπόν θα επιβληθεί αυτός ο φασισμός ε, μέσω του ψύχους, γι' αυτό αυτοί που αγαπούν την ελευθερία τελικά θα καταψηφίσουν αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Αμάλια Σαρτόρη έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον συνάδελφο Βιδάλ Κουάδρας για την έξοχη έκθεσή του και την έξοχη ικανότητά του διαμεσολάβησης που είναι κάτι αναγνωρισμένο που μας οδήγησε να ψηφίσουμε έναν κανονισμό που υποστηρίζεται ευρέω και μάλιστα στην πρώτη και μοναδική ανάγνωση. Και εγώ και η αντιπροσωπεία μου και η ομάδα μου με τα χαράς ψηφίζουμε αυτόν τον κανονισμό διότι σίγουρα είναι μια σημαντική πρόοδος, από τη σημαντική πρόοδος σε σχέση με τις παρελθούσες πολιτικές που ακολουθήθηκαν είναι ένα σημαντικό βήμα για μια μακρά διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσουμε όσον αφορά νέες και φιλόδοξες πολιτικές. Κάτι που ήδη ανακοινώθηκε από τον Επίτροπο. Είναι καλή αυτή η επιλογή που έγινε στο Κοινοβούλιο για μια πολιτική αλληλεγγύη όσον αφορά την εσωτερική αγορά που είναι και μια προειδοποίηση έναντι εκείνου που τα τελευταία χρόνια έπαιξε με αυτό τον τομέα. Θα πρέπει όμως να υπάρχουν διάφορες δίωδοι, οι να είναι πολλές και η ποιότητα να ελέγχεται των πηγών. Όσον αφορά αυτό, ίσως είναι πολύ μετριοπαθής η προσέγγιση που ακολουθήθηκε όσον αφορά τον νότιο διάδρομο. Συμφωνώ απόλυτα, συμμερίζομαι το ότι η αγορά είναι η μόνη εγγύηση για την καταπολέμηση των κινδύνων, κινδύνων που συνδέονται με τον εφοδιασμό. Όμως θα πρέπει να υπάρχει αγορά και θα πρέπει να εγγυηθούμε μία ανταγωνιστική αγορά, να ευνοήσουμε συνεπώς με κανόνες, με κανονισμούς, οδηγίες, χρηματοδοτήσεις, ε, πολλαπλά δίκτυα, πολλαπλές πηγές εφοδιασμού, ε, ούτως ώστε να μην υπάρχει πλέον μονοπόλιο στον τομέα. Ούτε όσον αφορά τις πηγές, ούτε όσον αφορά τα δίκτυα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία μου. Μάρικ Σίβιετς. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Ο ασφαλής εφοδιασμός σε φυσικό αέριο είναι ένα θέμα που είναι εξόχως στατηγικό Τέσσερι επιτροπέ επελήφθησαν του ζητήματο και τα επεξεργάστηκαν επιγόντω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αφορά γεωπολιτικά ζητήματα, τεχνολογικά θέματα, αλλά και το πνεύμα τη Ευρωπαϊκή αλληλεγγύης πάνω απ' όλα. Σε ποιο βαθμό θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εσωτερική αγορά σε αυτόν τον τομέα, σε ποιο βαθμό θα θέλαμε να κινηθούμε μέσα σε αλληλεγγύη, σε ποιο βαθμό οι ισχυροί μπορούν να προστατεύσουν τους αδύνατους έχει επιτευχθεί ένας συμβιβασμός, είναι κάτι που θα έπρεπε να μας χαροποιεί όπως κάθε συμβιβασμός, αλλά όταν θυμάμαι τις αρχικές μας φιλοδοξίες θέλω να προχωρήσουμε περισσότερο. Σαν σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο πιο σημαντικός, η πιο σημαντική λέξη για μας είναι ασφάλεια. Αλλά ασφάλεια των απλών ανθρώπων που πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, που διαβάζουν τις εφημερίδες και μαθαίνουν τις δυνατότητες που υπάρχουν να διακοπεί ο εφοδιασμό του φυσικού αερίου. Φοβούνται οι άνθρωποι ότι κάθε χειμώνα πρέπει να πληρώνουν περισσότερα και φοβούνται ότι δεν θα υπάρχει πλέον φυσικό αέριο. Ελπίζουμε αυτή η έκθεση τελικά να μειώσει, να καθησυχάσει του φόβου του. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ευθύ. Όταν ξεκινήσει η συζήτηση σχετικά με το πώ και ποιο θα καθορίζει τι απειλέ εναντίον του ασφαλού εφοδιασμού φυσικού αέριο, δεν υπήρξε συμφωνία. Προτάθηκε ότι μια απειλούμενη χώρα μπορεί να λάβει κάποια μέτρα. Ε, τώρα δύο χώρες και τώρα έχουμε αόριστους ορισμού σχετικά με αυτό. Αναφέρεται ότι κάποιοι φορείς θα ζητούν να ξεκινήσουν συζητήσει από αυτού του θέματο. Ένα μικρό βήμα, αλλά σημαντικό για την σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την δήλωσή σα. Επόμενο, κυρία Νικολά, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο θέματα. Την σημασία των χωρών παροχής φυσικού αερίου και των χωρών διαμετακόμισης. Θέλω να συγχαρώ φυσικά τον κύριο εισηγητή για τη στάση που κράτησε ενώπιον του προβλήματος αυτού. Εγώ είμαι εισηγήτρια για το Τουρκμενιστάν και πιστεύω ότι η χώρα αυτή μπορεί να παίξει ένα σημαντικό, ναζωτικό ρόλο ως χώρα τροφοδοσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των φυσικών πόρων τη και λόγω του ανοιχτού πνεύματο που έχει διατηρήσει εναντί τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε εξάλλου την δυναμικότητα που μπορεί να έχει η Κίνα στο μέλλον. Τα σχέδια αυτά, το Ναμπούκο, το Nord Stream κτλ. εξαρτώνται από τις σχέσεις μας με τις ε, χώρες παραγωγούς φυσικού αερίου που θα πρέπει να βασίζονται σε αμοιβαία παραδεκτά πρότυπα. <clears throat> Αν δεν έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση με τις χώρες αυτές, και να εξασφαλίσουμε με τον τρόπο αυτό και την πολιτική και την οικονομική σταθερότητα, δεν θα έχουμε τα πλεονεκτήματα τα οποία μπορούμε κατά τα άλλα να προσποριστούμε αν έχουμε αυτέ τι συμφωνίε. Και θέλω να πω ότι επίση ότι η χώρα μου, η Ρουμανία, έχει μια μεγάλη σημασία σαν χώρα διαμετακόμιση φυσικού αερίου. Πιστεύω λοιπόν ότι και η Ρουμανία και η Βουλγαρία μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για να εξασφαλίσουν την ενεργειακή σταθερότητα. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Μπιέλον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε η ασφάλεια εφοδιασμού σήμερα είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις της, εθνικής, της κυριαρχίας. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι έχει μία ενιαία φωνή μονάχα στα θέματα αυτά. Οι, πρόσφατες, οι κρίσεις του 2004 και 2005 και του 2008 κατέδειξαν τους κινδύνους της, επαρκούς ασφάλεια, της ανεπαρκούς ασφάλειας εφοδιασμού. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να προστατεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες της Κεντροανατολικής Ευρώπης από διακοπή εφοδιασμού στο φυσικό αέριο. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι έγινε κατά τη διάρκεια των δύο αυτών κρίσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας το 2008-2009. Καλύτερα να αντιδρούμε αργά παρά ποτέ. Πρέπει τελικά να κατανοήσουμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια κοινή ενεργειακή πολιτική και θα πρέπει να δημιουργήσουμε και τους απαραίτητους μηχανισμούς συντονισμού σε στιγμές κρίσης εφοδιασμού. Και φυσικά αυτό απαιτεί και μια ένα εξυγχρονισμό των διασυνδέσεων ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι ιδανική η συμβαστική λύση η οποία επετεύχθη Πιστεύω ότι αυτά τα οποία πρότεινε το Κοινοβούλιο καταρχήν ήταν πιο θετικά. Λαμβάνοντα όμω υπόψη όλα αυτά τα οποία είπα στην αρχή, πιστεύω πρέπει να υποστηριχθεί αυτή η πρόταση. Κοιτάξτε, ο ασφαλής εφοδιασμός, ο ενεργικός εφοδιασμός είναι ένα πρόβλημα που εμφανίστηκε στην κρίση φυσικού αερίου του περασμένου έτου. Η πρόταση περιέχει διάφορα μέτρα, ώστε να αυξηθεί ο ενεργειακό και η ασφάλεια για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά θέματα όμως ε, πρέπει να διευκρινιστούν. Έπρεπε να διευκρινιστούν και να βελτιωθούν. Στο Κοινοβούλιο έπρεπε να διευκρινιστεί ο ρόλος που μπορεί να διαδραματιστεί, τι γίνεται σε περίπτωση κατεπήγους ανάξης και πώς γίνεται, τι γίνεται με τις αμφίδρομες ροές, ε, τι γίνεται αναλογικότητα των δαπανών για συνοριακέ επενδύσει όσον αφορά τι υποδομέ. Διευκρινίστηκαν λοιπόν ε, οι όροι για να κηρυχθεί μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μέτρα μπορούν να λάβουν προληπτικά τα κράτη-μέλη, πώ τα προετοιμάζονται τα κράτη-μέλη μετά το Κοινοβούλιο έπρεπε να βελτιώσει την χρήση των ευαίσθητων πληροφοριών, ώστε να μην χρησιμοποιούνται με ε, ανεπίτρεπτο τρόπο. Όλα αυτά τα θέματα όμως τελικά παρέμειναν επίλυτα. Ο ορισμός των προστατευμένων χρηστών ε, και οι υποδομές ή τα πρότυπα για τις υποδομές ε, νη ένα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επεξεργαζόμαστε αυτά τα στοιχεία και μετά την έγκριση αυτού του κανονισμού. Σας ευχαριστώ. Ναι, ο Πρόεδρος, ε, σήμερα συζητάμε πιθανότατα ένα από τα σημαντικότερα έγγραφα ε, αυτή τη Ολομέλη, αυτή τη Συνόδου. Πολλοί πολίτε κατά τη διάρκεια του χειρότερου χειμώνα που πέρασαν το 2009 υπέφεραν. Υπέφεραν από το ψύχο. Ακραίε συνθήκε. Και εκεί διακόπη ο εφοδιασμό φυσικού στην Ευρώπη. Και εκεί βλέπουμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό ο κανονισμό αποδεικνύει ότι θέτουμε την ευμάρεια την, ε, και την άνεση των πολιτών πάνω απ' όλα. Αυτός ο κανονισμός τονίζει ότι όλα τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο του φυσικού αερίου θεωρούνται προστατευμένοι πελάτες. Ο κανονισμός αναφέρει επίσης ότι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν ούτως ώστε να, να παρέχονται επαρκείς ε, ποσότητε και σε ακραίε συνθήκε. Άρα χρειάζεται ενίσχυση των υποδομών στα διάφορα κράτη-μέλη, καθώ και οι διασυνδέσει μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε εύρυθμη λειτουργία των φυσικών βρόχων δηλαδή των αγωγών και των αναδρόμων ροών. Θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα λήψεως προληπτικών μέτρων για περιπτώσεις κρίσεω. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ζητήσει μια έγκαιρη εφαρμογή του κανονισμού ε, στα κράτη-μέλη. Χαίρομαι που ο εισηγητή έλαβε υπόψη διάφορα θέματα που απασχολούσαν τα κράτη-μέλη. Ο εισηγητή έλαβε υπόψη ε, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών μελών και ανάγκες τους. Οι προτινόμενες λύσεις είναι επαρκείς και για την Σλοβενία. Συνδεθήκαμε με τον αγωγό από την Αλγερία και νομίζω ότι έχουμε πετύχει τις αναγκαίες προδιαγραφές. Συγχαίρω επίσης τον εισηγητή, τον κύριο Βιδάλ Κουάδρας, ο με μεγάλη επιδεξιότητα διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Νομίζω ότι μας έδωσε ένα έξοχο κείμενο και ελπίζω να υποστηριχθεί αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Άννη Ποδηματά το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θέλω πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Βίνταλ Κουάντρα για τη σημαντική συμβολή του στην επίτευξη αυτού του περιεκτικού συνδυασμού με το Συμβούλιο και μάλιστα σε πρώτη ανάγνωση ο νέος κανονισμός έρχεται να αντιμετωπίσει σοβαρές εγγενείς αδυναμίες στην ασφάλεια εφοδιασμού της ένωσης με φυσικό αέριο με την ενίσχυση της δράσης των δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ευρωπαϊκού συντονιστικού οργάνου με τη θέσπιση κριτηρίων έγκαιρης προειδοποίησης και επαγρύπνησης και βεβαίως με τις ρήτρες προστασίας και καλύτερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών και ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πρέπει να αποτελούν τη βασική μας προτεραιότητα. θέλω ωστόσο να επισημάνω το τονίζει συνεχώς το κοινοβούλιο ότι χρειάζεται να υπερβούμε τις αποσπασματικές προσεγγίσεις στα θέματα της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και να προχωρήσουμε σε μια συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της ενέργειας με την ενίσχυση σε πρώτη φάση της περιφερειακής συνεργασίας και την προώθηση έργων διαφοροποίησης πηγών ε, και οδών εφοδιασμού όπως είναι ο ναμπούκο και ο itgi έργα συμπληρωματικά και όχι αντιπαραθετικά που μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην ασφάλεια εφοδιασμού της ένωσης. Σε ευχαριστώ πολύ. Ιβο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Πέρσι περάσαμε μια μεγάλη ενεργειακή κρίση, ήταν δυσάρεστη. Όμως δεν οφειλόταν σε διαθετικά προβλήματα της αγοράς, δομικά προβλήματα. Οποιαδήποτε προβλήματα ε, που εμφανίστηκαν ήταν περιτά. Θα πρέπει να αποφύγουμε στην επίλυση των προβλημάτων να αυξηθεί η τιμή που καταβάλει ο τελικός καταναλωτής. Πρέπει να προσέχουμε πολύ όταν ορίζουμε το ποιος είναι προστατευμένος πελάτης. Να μην είναι πολύ ευρύς ορισμός. Διαφορετικά η τελική τιμή του φυσικού αερίου θα αυξηθεί. Δεύτερον, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όσον αφορά τον ορισμό της ε, περίοδου της υποχρεωτικής κατά την οποία θα πρέπει να εξασφαλίζουν ασφαλή εφοδιασμό οι προμηθευτές. Να μην είναι 60 μέρες, να είναι 30 μέρες. Διαφορετικά θα πρέπει να δημιουργήσουμε τεράστιους χώρους αποθήκευσης και αυτό θα αντικατοπτήσει την τελική τιμή του φυσικού αερίου και χρειάζεται και πιο σαφής ε, ορισμός της ψυχροτέρας περίοδου. Ευχαριστώ επόμενος ομιλητής, ο κ. Μαρκίνβιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κ. Ματσινκίεβιτς μάλλον. Συγχαίρομαι τον εισηγητή μας, τον κύριο Αλέχο Βιδάλ Κουάδρας, που πριν από ένα χρόνο αντιμετώπισε μια πάρα πολύ σοβαρή κρίση να ετοιμάσει να ετοιμάσει μια έκθεση για το ασφαλή εφοδιασμό ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εργάστηκαν προς επίτευξη συμβιβασμού. Ο κανονισμός όσον αφορά τον ασφαλή εφοδιασμό σε φυσικό αέριο θα πρέπει να διευκολύνει τελικά τις δράσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να υποχρεώσει όλους τους φορείς να ε, δρούν βάσει της αρχής της πρόληψης. Όπως ακούσαμε από τον εισηγητή, μας είπε ότι το έγγραφο αυτό δίνει απαντήσεις ή προσπαθεί να δώσει απαντήσεις όσον αφορά τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η προσπαθει να δωσει απαντησει οσον αφορα τα Ένωση. Δεν θα σχολιάσω τη γενική κατάσταση και να πω ότι βεβαίω μπορεί να εμφανιστεί κάποια νέα κρίση κάποια στιγμή. Βλέπουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βλέπουμε και τι γίνεται και στις σχέσεις μεταξύ Πολωνίας και Ρωσίας όσον αφορά το θέμα αυτό. Μιλώ για τη Σύμβαση για το Φυσικό Αέριο. Και αυτή είναι μια νέα πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γίνεται πεδίο μάχης η Πολωνία, πεδίο μάχης μαχών μεταξύ τη Ρωσική Ομοσπονδία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την απελευθέρωση τη αγορά του φυσικού αερίου. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να τα καταφέρει καλά εδώ θα πρέπει να εστιαστεί στις, ε, στη διαφοροποίηση. Η Πολωνία είναι πολύ περιορισμένη όσον αφορά τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα μιας τεράστιας κρίσης όσον αφορά τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο και η πολωνική οικονομία ίσως να υποφέρει σοβαρά προβλήματα, να υποστεί σοβαρά προβλήματα. Και βασιζόμαστε στην υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να είναι στο πλευρό μας Είμαστε μια χώρα διαμετακόμισης, διέλευσης. Δεν είμαστε τελικός προορισμός όσον αφορά το δρόμο μεταφοράς του φυσικού αερίου και ελπίζω όλα τα κράτη-μέλη να εκτιμήσουν τη δράση που πρέπει να αναλυθεί όσον αφορά την ασφάλεια σε φυσικού, σε φυσικό αερίο. Κύριος Χούτας. Κύριος Χούτας, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέψει τον εαυτό της να εξαρτάται από εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας φυσικού αερίου που να μην είναι ασφαλή. Η κρίση του 2009 μας κατέδειξε ότι είμαστε ιδιαίτερα ευάλωτοι γιατί δεν έχουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή κοινή στρατηγική στον τομέα της ενέργειας. Οι συνέπειες αυτές της κρίσης ήταν απτές στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως στους στρωτού και ευάλωτους καταναλωτές. Κατέδειξε λοιπόν σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη είναι αλληλένδετα στην εξάρτησή του από φυσικό αέριο. Είναι απαραίτητο λοιπόν ω εκ τούτου να αναπτύξουμε μια στρατηγική η οποία θα διαφοροποιήσει τις οδού ε, τροφοδοσίας και παροχής φυσικού αερίου και να αποκτήσουμε και μια ικανότητα αντιμετώπισης παρομοίων κρίσεων. Βάσει της συνθήκης Λισαβόνας είναι απαραίτητο να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός τροφοδοσίας για το φυσικό αέριο. Το σχέδιο Ναμπούκο μέσα στα πλαίσια του μηχανισμού έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα μια ιδιαίτερη σημασία. Θα πρέπει να υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή τη στιγμή είναι η μόνη εναλλακτική λύση για το ρωσικό μονοπόλιο. Το λόγο τώρα για ένα λεπτό Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο εισηγητής κατάφερε να πετύχει ένα συμβιβασμό ιδιαίτερα δύσκολο πρέπει να πω. Τον ευχαριστούμε λοιπόν. Τον ευχαριστούμε γιατί δεσμεύτηκε και βοήθησε σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ ακόμη κύριε Επίτροπε που ασχοληθήκατε με το θέμα της Πολωνίας και της Ρωσίας. Η ενέργεια είναι συντελεστής κλειδί στην Ευρώπη. Ε, εξαρτάται η ανεξαρτησία μιας χώρας. Κάποιοι μέσα σε αυτή την αίθουσα μιλήσανε ε, σαν να ήταν η ενέργεια μόνο οικονομικό ζήτημα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πολλές χώρες στην Ευρώπη θεωρούν την ενέργεια συντελεστή ανεξαρτησίας. Για να πιστείτε δεν έχετε παρά να στραφείτε προς τη Ρωσία. Η Ρωσία παίζει σε δύο γήπεδα. Παίζει στο οικονομικό γήπεδο, αλλά παίζει και στο πολιτικό. Και το θέμα της ασφάλειας. Αυτό που μας λείπει σήμερα είναι μια μεγαλύτερη δέσμευση εκ μέρους των φορέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας έδινε τη δυνατότητα να παίξουμε και εμείς σε δύο γήπεδα σε αυτό το ζήτημα. Κυρία Τόγια. Α, ε, I'm sorry. Ε, το... Πρώτα για 1,5 λεπτό ο κύριος Γιούρκ. Και μετά κυρία Τόγια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με εκείνους τους ομιλητές που είπαν ότι η πρόταση για κανονισμό όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού είναι καλός τρόπος για να προστατευτούμε από κρίσεις στο μέλλον. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε τη διάταξη των προστατευμένων πελατών. Τώρα μιλάμε και για τις μικρές επιχειρήσεις που θα έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση και προστασία. Δεν μιλάμε για μικρό αριθμό πολλατών σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για την Ουγγαρία παραδείγματος χάρη 600.000 νοικοκυριά και η προστασία των μικρών επιχειρήσεων μας έδειξε το 2009 ότι μπορεί να χρεοκοπήσουν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις όταν υπάρχει διαταραχή εφοδιασμού. Σας υπενθυμίζω ακόμη ότι ο κανονισμός αυτός και η έγκρισή του θα είναι σημαντικό βήμα, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις επίγουσες ανάγκες επενδύσεων που έχουμε. Τέσσερα κράτη-μέλη στείλανε την περασμένη εβδομάδα μια επιστολή στον Επίτροπο Ενέργειας για να ζητώντας να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα ώστε να υπάρξει και σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό των 7 ετή. Η εξασφάλιση εφοδιασμού ενεργειακών πηγών σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε τα δίκτυα και αυτό πρέπει να αντανακλάται στον προϋπολογισμό. Η επόμενη εγγεγραμμένη ομιλήτρια δεν φαίνεται να είναι στην αίθουσα, οπότε το λόγο θα πάρει η κυρία Κορχόλα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Βίδαλ Κουάδρας για την ε, μεγάλη υψηλή ποιότητα της εκθέσεώς του. Πόσο φυσικό αέριο θα πάρουμε ήδη πρέπει να το εξασφαλίσουμε από τη Ρωσία και θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ευρωπαϊκή υποδομή η οποία θα εξασφαλίσει τη σωστή ροή του αερίου και να αντιμετωπίσει καταστάσεις κρίσεως. Θα πρέπει να αναλάβουμε λοιπόν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει η ασφάλεια. Τροφοδοσία σε φυσικό αέριο. Η ιστορία και το παρελθόν μας δείχνει πόσο απαραίτητο είναι κάτι τέτοιο. Σήμερα είμαστε ακόμα σε κατάσταση ε, επικίνδυνης εξάρτησης. Πάνω από το 30% του φυσικού αερίου της Ευρώπης είναι εισαγόμενο και αυτή η εξάρτηση μπορεί να ανέβει σε μερικά χρόνια πάνω από το 50% μέχρι και το 70%. Θα μπορούσε όμως βοηθήσει το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, και η αποθήκευσή του. Αυτό όμως απαιτεί νέες υποδομές. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη διανομή φυσικού αερίου και καλύτερη ασφάλεια του εφοδιασμού. Επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις δυνατότητε των ανανεώσιμων ενεργειών. Ούτω ή άλλω, η κρίση μεταξύ τη Ρωσία και των ομόρων αυτή τη χώρα έδειξαν πόσο εξαρτώμεθα από τη χώρα αυτή για την τροφοδοσία μα σε φυσικό αέριο. Ω εκ τούτου, θα πρέπει να, εξαρτη... να έχουμε στο μυαλό μα την αρχή τη ε, αλληλεγγύη στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίση και για τι χώρε, οι οποίε είναι όμορε τη Ρωσία, Θα πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτέ. για ένα λεπτό παρακαλώ. Ačiū, gerima pirmininkė, gerimas komisarė, kolegos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τιμήσω τα μέλη του Κοινοβουλίου που συνέταξαν αυτή την έκθεση. Η αυξανόμενη εξάρτησή μας από τους προμηθευτές ενέργειας τρίτων χωρών είναι μια νέα πολιτική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συντονίσουμε τις προσπάθειες μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Πρέπει να εργαστούμε όχι μόνο σε περιόδους κρίσης αλλά κυρίως όταν συντάσσουμε τις πολιτικές της Ευρώπης στον ενεργειακό τομέα και κυρίως όταν προσχωρούμε σε συμβάσεις με τρίτα μέρη. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ζητήσω ε, όταν συνταχθεί ε, η σύμβαση για μάλα με τη Ρωσία, παρακαλώ, να μην δημιουργήσει αρνητικό προηγούμενο για το μέλλον. Μόνο η ελληνική θα μπορέσει να μας εξασφαλίσει ασφαλή εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ διαδικασία Catch the Eye. Έχουν ζητήσει το λόγο αρκετοί συνάδελφοι για αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Κέλαμ. Σας παρακαλώ πολύ ένα λεπτό για να μπορέσουν να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Κύριε Κέλαμ, you have the floor. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει ότι η Ευρώπη έχει πάρει πλέον το ουσιαστικό μήνυμα από τις πολλές κρίσεις. Η πρώτη εμπειρία της Εστονίας ήρθε το 1992 όταν η Ρωσία έκλεισε όλη την παροχή αερίου και πετρελαίου. Αλλά αυτό μας ενδυνάμωσε πρέπει να σας πω. Σήμερα όμως βλέπουμε θετική συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Έτιγκερ για την υπεύθυνη προσέγγιση που υιοθέτησε για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων πρέπει να εντάξουμε την αλληλεγγύη στους πρακτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι θα δημιουργήσουμε κοινά πρότυπα υποδομής και εφοδιασμού θα ενισχυθεί ο συντονισμός από την Κομισιόν αλλά κυρίως αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ολοκληρωμένο δίκτυο εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνομαι στο, την πρόταση Τούρμες να βελτιωθεί η διασύνδεση μεταξύ Βορρά και Νότου και να αποκτήσουμε και αποθηκευτικούς χώρους για το μέλλον. Είναι σωστή η πρόταση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί σαν κοινότητα όταν προασπιζόμαστε τα ενεργειακά μας συμφέροντα και πρέπει και τα κράτη-μέλη να είναι ενεργά ιδιαίτερα εκείνα που δεν έχουν λύσει τις διμερείς τους σχέσεις με τη Ρωσία. Η Ουγγαρία έχει εισαγωγές για το αέριο και 80% προέρχονται από τη Ρωσία. Συνεπώς η εξάρτηση των οικοκυριών μας είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ιδιαίτερα όταν μιλάτε για τα νοικοκυριά κυριά που χρησιμοποιούν περιφερειακή διανομή και γι' αυτό θα θέλαμε να διαφοροποιήσουμε τις ενεργειακές πηγές και τα δίκτυα διανομής. Υποστηρίζουμε λοιπόν 100% τη δημιουργία του Ναμπούκο και άλλων αγωγών και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι πραγματικά χρησιμοποιούμε όλους τις ε, τους κοινοτικούς πόρους προς αυτή την, κατεύθυνση. Βεβαίω το φθηνότερο για μας θα ήταν εφοδιασμός από την Ουκρανία. Σταθερός εφοδιασμός όμως. Γι' αυτό θα ζητώ από τον Επίτροπο να λειτουργήσει κοινοτικά ώστε να ρυθμίσει τα πράγματα με τη Ρωσία και την Ουκρανία και να υπάρχει και ένα σύστημα εγγύησης ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Για την κυρία Τόγια δεν τη βλέπω στην αίθουσα, οπότε το λόγο θα πάρει ο κύριος Μπούτικοφέρ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Έτιγκερ σε σχέση με δύο σημεία τα οποία ανέφεραν προηγουμένως οι συνάδελφοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τούρμες αναφέρθηκε ιδιαίτερα σαφώς στο θέμα της ικανότητας πρόβλεψης της ζήτησης σε φυσικό αερίο. Εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία στην παροχή αερίου, τον εφοδιασμό, αλλά αυτό είναι μονάχα η μία πλευρά του νομίσματος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε πώς εσείς μπορείτε να έχετε προβλέψεις για το μέλλον για να μπορείτε να δείτε και την άλλη πλευρά, την πλευρά της συζήτησης και να την ενσωματώσετε στη στρατηγική μας. Δεύτερον, επανερχόμαι σε αυτά που είπε ο κ. Σφόμποντα. Θα ήθελα να σκεφτούμε περισσότερο για την κοινότητα ενέργειας στην ευρωπαϊκή ενέργεια. Υπάρχει η δεξαμενή σκέψη με επικεφαλή στον κύριο Ντελόρ που έχει αντιμετωπίσει το θέμα αυτό αλλά για σας είναι αυτό ένα θετικό βήμα, μια θετική κίνηση που διατρέχει και το έργο σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στη συζήτηση αυτή για την ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ θα ανατονίσω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μεγαλύτερη διαφοροποίηση για την παροχή φυσικού αερίου σε παγκοσμίο επίπεδο. Αλλά αυτό το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό σε σχέση με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κρίση του πετρελαίου που θα αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει με ενεργό τρόπο την ε, αντικατάσταση των ε, πηγών του πετρελαίου που ήδη δηλείστε στα σύνορά της με φυσικό αέριο. Αλλά φυσικού αερίου που προέρχεται από μη <clears throat> ε, ορυκτά, ορυκτές πηγές, αλλά που παράγεται αντίθετα από καύση απορριμμάτων όπως γίνεται στην Ελβετία, όπως γίνεται στην ε, Σουηδία και στην Ισπανία. Αυτός είναι ένας τρόπος παραγωγής φυσικού αερίου που πρέπει να προωθηθεί με επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα παρόν στις σκέψεις μας όταν αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή επάρκεια. Die meisten Gasanbieter haben aufgrund οι περισσότεροι καταναλωτές ε, φυσικού αερίου έχουν μια αυξανόμενη ζήτηση η οποία οδηγεί και σε αυξανόμενο τίμημα ενέργειας. Η Μόσχα μπορεί να αντιμετωπίσει και τον επόμενο χειμώνα πάλι κρίση τροφοδοσίες σε φυσικό αέριο. Τα μέτρα τα οποία λάβαμε το χειμώνα ήταν ε, κατόπιν εορτής. Είναι απαραίτητο να έχουμε ταχύτερες δυνατότητες ε, αντίδρασης όταν έχουμε και μια νέα κρίση. Επομένως θα πρέπει να δώσουμε μια μεγαλύτερη προσοχή στην κρίση, ε, στην αντιμετώπιση των κρίσεων και επίσης θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα ε, εργοστάσια παραγωγής με ποινική ενέργεια στη Γερμανία και στις μονάδες ε, ρευστοποίησης του άνθρακα πριν από την καύση του, όπως είναι στην Πολωνία. Η κρίση αυτή μας έδειξε ότι το ευρωπαϊκό σύστημα τη ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τι δυνατότητε που του παρέχει η συνθήκη Λισαβόνα ώστε να μην είμαστε εξαρτημένοι από τη Ρωσία. Ακόμα και το σχέδιο Ναμπούκο δεν θα λύσει το πρόβλημα τη εξάρτηση. Θα πάρει για ένα λεπτό πάλι ο κύριο Γκρίζερ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, ο Επίτροπος μας είπε ότι πρόκειται για το πρώτο κείμενο μετά τη Λισαβόνα για το τομέα της ενέργειας και περιλαμβάνει την αρχή ενεργειακής ε, αλληλεγγύης. Επανέρχομαι στη χώρα μου, την Πολωνία. Η κρίση του 2009 αλλά και οι προηγούμενες κατέδειξαν ότι χωρίς ενεργειακή αγορά, χωρίς υποδομές, χωρίς διασυνδέσεις, ο συντονιστικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς πολιτική θέληση εκ μέρους της Επιτροπής και του Συμβουλίου δεν μας δίνει τη δυνατότητα να επιλύσουμε αυτές τις κρίσεις. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή η Πολωνία, πρέπει να σας πω, έχει μια συμφωνία για 2,5 εκατομμύρια κυβικά η κατάσταση θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, ιδιαίτερα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ρόλο του είπα του εκπροσώπου εξωτερικής πολιτικής. Ο Επίτροπος Αττικέρ μας λέει ότι σε δύο-τρία χρόνια θα πρέπει να ανασκοπήσουμε αυτό το κείμενο για να δούμε σε ποιο βαθμό είναι αποτελεσματικό. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία από τώρα. Ευχαριστώ ε, Securitatea energetică a Uniunii Europene depinde de diversificarea... Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από τη διαφοροποίηση των πηγών και των αγωγών. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην υποδομή και στην αποτελεσματικότητα της χρήσης της ενέργειας. Όσον αφορά λοιπόν την υποδομή των αγωγών, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε νέους αγωγούς Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικός ο Ναμπούκο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη πρέπει να επενδύσει περισσότερο για την αποθήκευση του αερίου και να, να επενδύσει και για τη βελτίωση των διασυνδέσεων μεταξύ κρατών μελών. Όλες αυτές οι διασυνδέσεις πρέπει να δημιουργηθούν όπου υπάρχει η ανάδρομη ροή. Δεν πρέπει όμως και να ξεχνάμε τις ανανεώσιμες πηγές. Βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας έχουμε ένα νέο πλαίσιο συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης και νομίζω ότι ο εισηγητής Βιντάλ Κουάντρας είναι άξιος συγχαρητηρίων γιατί αυτός ο κανονισμός είναι ένα βήμα προς τα πρόσωπα όσον αφορά την ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βιντάλ Κουάντρας και τον Επίτροπο Εωτίνγκερ. Σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι αυτό το τόσο σημαντικό νομοθέτημα έχει συνταχθεί και είναι τώρα έτοιμο για έγκριση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες εξατώνται από τις ρωσικές εισαγωγές ε, φυσικού αερίου κατά 100%. Αυτή είναι μια κατάσταση μεγάλης εξάρτησης και μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική εκμετάλλευση. Αυτό είναι λοιπόν πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να προχωρήσουμε προς μορφές ενέργειας που ελαχιστοποιούν την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακο και επίση θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο έκτακτη ανάγκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να έχουμε τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση πραγματική κρίση. Τα στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν στην έκθεση αυτή είναι και το σύνολο περίπου του, της κατανάλωσης μιας χώρας όπως η Σλοβακία πρέπει η ασφα... σε φυσικό αέριο να λειτουργεί απρόσκοπτα και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλείας σε κρίση και από θέματα ασφαλείας. Γι' το πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι μια μεγάλη συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων αυτών. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Έτιγκερ. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Βιντάλ Κάντρας για την πολύ σημαντική του έκθεση. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο εφοδιασμός ο ενεργειακός για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός. Ε, δεν ακούμε τον ομιλητή, ε, το μικρόφωνο έκλεισε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές εφοδιασμού για το αέριο και να βρούμε ε, τις πολιτικές λύσεις και τις οικονομικές τις πιο επωφελείς. Το κλειδί της ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει από τη βελτίωση της υποδομής των διασυνδέσεων και από τη δυνατότητα ανάδρομης ροής και πρέπει να, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να παρακολουθήσουμε τα πράγματα με πνεύμα αλληλεγγύης. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν τις συζητήσεις για την κοινότητα την ενεργειακή. Ε, ήσασταν και σύντομος. Η κυρία Γιαρζεβιέκα έχει το λόγο παρακαλώ. Ο κύριος, ο κύριος, ε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο κύριος Τζα... Τζαρζοβιέκα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Α, κυρία, με συγχωρείτε, ήταν λάθος. Yes, I'm sorry. Dziękuję. Rozporządzenie, które dziś przegłosujemy, jest krokiem milowym w budowaniu. Η έκθεση που θα ψηφίσουμε σήμερα είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου στην ενεργειακή πολιτική. Έχουμε ακούσει όλες τις εκκλήσεις για αλληλεγγύη που θα οδηγήσουν σωστή και ομαλή λειτουργία των νομοθετικών μέσων για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε γρήγορα σε περίπτωση κρίσης. Το κείμενο που θα ψηφίσουμε αργότερα ε, βέβαια ξεφεύγει κάπως από τη φιλόδοξη προοπτική που είχε το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά υπάρχει κάποιος μηχανισμός για τη διαχείριση της κρίσης. Το γεγονός ότι μπορέσαμε να βρούμε μια γρήγορη συμφωνία με το Συμβούλιο είναι θετικό μήνυμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, κύριο Βιντάλ Κουάντρας, που ήταν ανοιχτός με προτάσεις εξ αρχής ανοιχτός στις σκέψεις των συναδέλφων και χάρη στο συμβιβαστικό του πνεύμα μπορέσαμε να οδηγηθούμε σε ένα κείμενο που γίνεται αποδεκτό από όλους. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι ε, όργανο κλειδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αγωνιστούμε για φιλόδοξα μέτρα που καμιά φορά μοιάζουν ανέφικτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και το Συμβούλιο και την Κομισιόν για τη συνεργασία του με το Κοινοβούλιο στα, θέματα, στα πλαίσια αυτού του νομοθετήματο. Είναι σαφέ ότι η νομοθεσία φυσικά είναι απλώ το προαπαιτούμενο για να υπάρξουν οι απαραίτητε επενδύσει. Χρειαζόμαστε τι ευρωπαϊκέ επενδύσει. Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε τι υποδομέ οι οποίε είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη κρίση για το μέλλον. Το νομοθέτημα αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι είναι απαραίτητη η αλληλεγγύη μεταξύ μα, είναι απαραίτητη η συνεργασία μα, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού για του πολίτε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ουγγαρία έχουμε πολλέ συζητήσει για τα αισθήματα αυτά και εμεί ω σοσιαλιστέ στην Ουγγαρία θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια εφοδιασμού στην ε, Ευρώπη. Αλλά ο επικεφαλή κυβέρνηση τη ε, Ουγγαρία τόνισε επίση ότι η Ουγγαρία θέλει να έχει απόλυτη απεξάρτηση από εξωτερικού φορεί ενέργεια και ελπίζουμε ότι αυτό θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα στο μέλλον. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Από το 2006 έγινε η πρώτη διακοπή εφοδιασμού από τη Ρωσία. Έκτοτε, ασφαλής εφοδιασμός ενέργεια έχει τη σημασία για τις δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά πολύ πολιτικό διότι έχει σοβαρές συνέπειε για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς και για τη διεθνή της θέση. Παρά το γεγονός ότι αυτό έχει αναγνωριστεί ευρέως, στην πράξη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανίκανη να σταματήσει την αυξανόμενη εξάρτησή τη από τον εφοδιασμό από διάφορου φορείς που έχουν πολιτικό πρόγραμμα και δεν διστάζουν να εκμεταλλευτούν την αυξανόμενη ευαλωτότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό οφείλεται στην αντίσταση κάποιων σημαντικών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όμως, για να κλείσω, θα ήταν εσφαλμένο να πούμε ότι δεν υπάρχει σύστημα ασφαλού ενεργειακού φωτισμού τώρα υπάρχει. Μόνο που είναι κατακαιρματισμένο και όχι συλλογικό. Κάθε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ενώση θέλει να προστατεύσει τον εαυτό τη μέσω των σχέσεων με του διαφόρου ε, προμηθευτέ και κάνουν και ανταγωνισμό για να του προσελκύσουν. Λόγο στην κυρία Τζαβέλα για μια σύντομη παρέμβαση, γιατί έχει ήδη λάβει μέρο στη συζήτηση. Κυρία Πρόεδρος, επειδή αρκετοί από εμά σε αυτή την αίθουσα αναφερθήκαμε στο Ναμπούκο ως ένα πολύ σημαντικό έργο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Επίτροπο αν μπορεί να μας πει πού βρίσκεται το έργο αυτό και τι έχει προχωρήσει ως προς το θέμα του Ναμπούκο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτροπε, θα κλείστε εσείς τη συζήτηση. Ο εισηγητής δεν προβλέπεται να παρέμβει πάλι. Εξάλλου, κύριε Βιντάλκου Άντρα, πράξατε την αποδοχή των θέσεών σας από τους συναδέλφους. Mr. Commissioner, you have the floor. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η συζήτηση που έλαβε χώρα ήταν εξαιρετική. Νομίζω ότι έχουμε δώσει και μια μεγάλη όθηση στην ενεργειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά εξαρτώμεθα από το φυσικό αέριο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα της ε, έλλειψης μελλοντικά του πετρελαίου και του άνθρακα από την, από την διεθνή αγορά και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλο και περισσότερο τις ε, ανανεώσιμες ενέργειες για να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της Ευρώπης. Επίσης, στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητος, που είναι ένας από τους σημαντικούς μας στόχους, θα πρέπει να μην σπαταλούμε ενέργεια, αλλά να τη χρησιμοποιούμε επωφελώς. Θέλουμε λοιπόν μέσα στους επόμενους μήνες να συζητήσουμε αυτό το θέμα μαζί σας και να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα. Αναφέρθηκε επίσης η κοινότητα ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λειτουργήσει σε μια κοινότητα που είναι όλο και πιο αλληλέγγυα και πιο επωφελή. Αυτή είναι και η κατεύθυνση που έχει δώσει η ομάδα του κυρίου Ντελόρ. Εμείς θέλουμε στα επόμενα χρόνια να χρησιμοποιήσουμε τα νέα εργαλεία που μας δίνει το άρθρο 94 της Συνθήκης της Λισαβόνας με δυναμικό τρόπο ως νομική βάση ώστε να λάβουμε τα απαραίτητα ε, μέτρα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής ενέργειας γιατί δεν έχουμε ακόμα εσωτερική αγορά πλήρη σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στα χέρια ακόμα των κρατών μελών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μιλάνε για για κοινή πολιτική ενέργειας το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, αλλά στη συνέχεια κοιτάνε μονάχα τι δικές τους ανάγκες και την ανάγκη της δικής του βιομηχανία στα κράτη-μέλη. Είναι απαραίτητο λοιπόν να προχωρήσουμε με τα κράτη-μέλη για μια βελτίωση της κατάστασης επί τη βάση των νέων νομικών βάσεων. Και χώρες όμορες όπω είναι η Σερβία, η Κροατία, η Νορβηγία, χώρε ακόμα όπως και το Μαρόκο, οι χώρες του Μαγκρέπ, η Μέση Ανατολή, η Μολδαβία, η Ουκρανία, όλες αυτές οι χώρες είναι πραγματικοί εταίροι οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και η Τουρκία επίσης σε μια ευρύτερη ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου ζητήθηκε να προβλέψω ποια θα είναι η εξέλιξη της ζήτηση στην αγορά φυσικού αερίου. Εμείς θα παρουσιάσουμε προβλέψεις μέσα στον οδικό χάρτη για τα θέματα ενεργείας και αυτό θα περιλαμβάνει και την ε, Βέβαια, συγγνώμη, ε, τα κράτη-μέλη έχουν ακόμα την επιλογή του ενεργειακού μείγματο. Είναι τα κράτη-μέλη τα οποία αποφασίζουν πόσο φυσικό αέριο, πόσο πετρέλαιο και πόσο άνθρακα θα χρησιμοποιήσουν. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κάνει τις προβλέψεις και τις προτάσεις για το μέλλον γιατί αυτή θα πρέπει να είναι η βάση της ενεργειακής πολιτικής. Εμείς ξέρουμε ότι θα χρειαστούμε πάνω από 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου Μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 6 δισεκατομμύρια ή μπορεί να μειωθούν και σε 3 δισεκατομμύρια, αλλά το ερώτημα είναι να έχουμε την απαραίτητη υποδομή για να αποτρέψουμε μια εξάρτηση στο μέλλον. Και τονίζω και πάλι το θέμα της ανεξαρτίας. Θα πρέπει της ανεξαρτησίας στον εφοδιασμό. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια αξιόλογη αντιμετώπιση στον τομέα αυτό. Είναι γεγονός αυτό που είπατε ότι σε καταρχήν κατά 25% της ευρωπαϊκής τροφοδοσίας με φυσικό αέριο ότι προέρχεται από τη Ρωσία. Είναι πολύ. Ένα τέταρτο λοιπόν είναι η τροφοδοσία από την Ρωσία. Αλλά φυσικά χώρες όπως η Λετωνία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Βουλγαρία έχουν πολύ μεγαλύτερη ποσοστία εξάρτηση, πάνω από 50% άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία μηδενική εξάρτηση. Αυτό εξαρτάται από την γεωγραφική θέση της κάθε χώρας και από την απόσταση που έχει από τον τροφοδότη σε φυσικό αέριο, δηλαδή τη Ρωσία στην περίπτωση αυτή. Έχουμε επίσης όμως φυσικό αέριο από την Νορβηγία και την Αλγερία και θέλουμε να δώσουμε και μεγαλύτερη έμφαση στην τροφοδοσία με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη Μέση Ανατολή, το Κατάρ κτλ. Όλα αυτά λοιπόν θα μας οδηγήσουν σε αυξημένη ανεξαρτησία έναντι της Ρωσίας. Πρέπει να δούμε τα θέματα αυτά σε επίπεδο εταίρου. Είχαμε αναπτύξει ήδη από πέρσι τον ενεργειακό διάλογο μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Είναι αμφίδρομη λοιπόν αυτή η σχέση. Γιατί θα πρέπει να υπάρξει και χρηματοδότηση από τη Ρωσία για τον διάδρομο Nord Stream. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει η ροή φυσικού αερίου και στο μέλλον η Ρώση μπορεί να χρειαστεί να αγοράσουν προϊόντα βιομηχανικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τεχνογνωσία από την Ευρώπη για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της ρωσικής οικονομίας μέσα από την πώληση φυσικού αερίου. Δηλαδή αν έχουμε λοιπόν ε, έμφαση σε μία <clears throat> αμοιβαία εξάρτηση και όχι απλώς τη δυνατότητα η μία πλευρά να εκβιάσει την άλλη θα μπορούν να είναι επωφελείς η εταιρική μας σχέση με την ε, Ρωσία. Επίση, στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουμε την απαραίτητη ανάπτυξη υποδομών ώστε να μην μα περιορίζουν οι τεχνικέ ε, δυνατότητε. Και οι Ρώσοι, τονίζω και πάλι, θα πρέπει να είναι οι εταίροι μας στα πλαίσια της ε, ε, εμπορίας του φυσικού αερίου και Εξάλλου έχουμε τις εναλλακτικέ δυνατότητες από την Κασπία. Η Κασπία είναι το μεγαλύτερο, έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο και θα πρέπει με τη συνεργασία των Ρώσων να έχουμε τη δυνατότητα οι Ρώσοι να διαμετακομίσουν και φυσικό αέριο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν οι άλλε πηγέ, όπω είναι τη Νορβηγία και τη Αλγερία, που δεν εξαρτώνται από τη Ρωσία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα εξασφαλίζει ότι η τροφοδοσία μας θα γίνεται με το συντομότερο τρόπο από την Κασπία χωρίς να περνάει κατά από τον έλεγχο των Ρώσων. Αυτό προϋποθέτει όμως και μια αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θέλω να ζητήσω από όλα τα κράτη-μέλη, από την Ουγγαρία ως την ε, Ρουμανία και τη Βουλγαρία και την ε, Αυστρία, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την διαθεσιμότητα να δώσουμε μια λύση στα θέματα του νοτίου διαδρόμου του Ναμπούκο που θα εξασφαλίσει και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι αποφασιστικό. Εάν λοιπόν δεν παρασυρθούμε από προτάσεις οι οποίες δεν ευνοούν την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουν γίνει συναντήσεις για το Ναμπούκο. 1η Οκτωβρίου θα γίνει μια συνάντηση κορυφή και με το Τουρκμενιστάν. Αλλά οι αποφάσει δεν περιλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνονται από του επενδυτέ μεν. Πρέπει όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι είναι το δυνατόν, ώστε χώρε όμορε και χώρε παραγωγή, όπω είναι το Αζερβαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν, να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτό το σχέδιο και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό το να μπορεί να τεθεί στην σωστή κατεύθυνση. Και φυσικά στη συνέχεια, όπω είπατε, θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσει. Εγώ σα. Ε, υπόσχομαι ότι κάθε ευρώ το οποίο μπαίνει από τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την χρηματοδότηση αυτών των υποδομών θα χρησιμοποιηθεί εποφελώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές είναι μια σειρά αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν στο ορατό μέλλον. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν οι αποφάσεις αυτές και αν χρειάζονται περισσότερα χρήματα θα πρέπει και τα κατημέλη και το Κοινοβούλιο να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες. Φυσικά θέλω να ακούσω και την απόψη του Κοινοβουλίου για όλα αυτά τα ζητήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την έμφαση που δώσατε στο θέμα αυτό και ελπίζω ότι θα μπορέσει ο κανονισμός αυτός να εγκριθεί και να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατό και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε την αγορά φυσικού αερίου και φυσικά μπορούμε να έχουμε και μια διεύνηση του περιεχομένου αυτού του κανονισμού εκεί όπου αυτό είναι χρήσιμο και επωφελές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Έληξε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει στη συνέχεια. Και τώρα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι οι δηλώσεις